για τον προπολογισμό 2016. Εντολή για τον τριμερή διάλογο. Και καταρχάς για τέσσερα λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαιρετώ την Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Γεώργιαβα και όλου του συναδέλφου. Να θυμίσω ότι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μικρό προπολογισμό 1% του εθνικού εισοδήματος, 60 δις ευρώ σε πληρωμές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαρκώς αυξάνει τις αρμοδιότητές της και έχει διευρύνει και τη σύνθεσή της ως προς τα κράτη-μέλη. Ο προπολογισμό της που αν συγκριθεί με αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών σε ποσοστό του ΑΕΠ, στις Ηνωμένε Πολιτείες έχουμε το 20% του ΑΕΠ αλλά ε, ο δικός μας προπολογισμό έχει αυξημένη ε, ποιότητα και το 90% αφιερώνεται στην έρευνα. Μόνο 6% αφορά διοικητικές δαπάνες ή λειτουργίας. Είναι ένας προπολογισμό που εκπροσωπεί για πολλά κράτη-μέλη περισσότερο από το 50% των ε, επενδύσεων ως το 2016 θα πρέπει να καθορίσουμε τις προτεραιότητές μας που είναι τα τρία S, η απασχόληση, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Θα πρέπει λοιπόν μεταξύ άλλων να φροντίσουμε για την πρωτοβουλία των νέων, να φροντίσουμε για το 2014 και 2015, να ε, δούμε τι δεν πήγε καλά και για το 2016 το πρόγραμμα να πετύχει, να, να είναι σωστή πρικοδότηση του προγράμματος αυτού. Το προγράμματα όπως ο κόσμο, το κόσμο, η Ευρώπη του 2020 ή ο μηχανισμός για την διασύνδεση της Ευρώπης θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερη προσοχή. Όμως να μην ξεχνάμε και την εσωτερική αλληλεγγύη. Στην εσωτερική αλληλεγγύη έχουμε την πολιτική της συνοχή, η οποία επίσης βοηθά την ε, ε, ε, απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και την έρευνα. Πέραν του στόχου αυτού, θα πρέπει να μην ξεχνάμε και ένα στόχο αυτών της αλληλεγγύης, της στήριξης των φτωχότερων, των κρατών με τις μεγαλύτερες δυσχέρειες. Την κοινωνική διάσταση για τους πολίτες, την εσωτερική δηλαδή διάσταση που και για μας είναι προτεραιότητα. Και στην εξωτερική αλληλεγγύη όμως μας απασχολεί τι γίνεται στην Ουκρανία, τη Συρία, στην Μεσόγειο Υπ' αυτήν την έννοια, το κεφάλαιο 3 και το κεφάλαιο 4 είναι για μας πολύ σημαντικά. Και επίσης επαναλαμβάνουμε ότι οι περικοπές που γίνονται στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς δεν μπορεί να είναι περικοπές που θα κάνουμε αβίαστα ε, χωρίς να το ξανασκεφτούμε. Πρέπει να σκεφτούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, το κόστος που θα έχουν αυτές οι περικοπές. Η δημοσιονομική παρακολούθηση λόγω χάρη είναι σημαντική γιατί οργανισμοί όπως αυτό για τη μετανάστευση έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστος από ότι οι δαπάνες που απαιτούν. Θα πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε τις υποσχέσεις μας, να σεβαστούμε το πλαίσιο που έχουμε ορίσει για τις πληρωμές, να σεβαστούμε τις προτεραιότητες του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, την ευελιξία που θέλουμε και ελπίζουμε στο μέλλον το ε, Συμβούλιο να τηρήσει μια στάση σεβασμού των ε, υποσχέσεων, τις αναγγελίες και ανακοινώσεις που έχει κάνει, να τις μεταφράσει ως άρκα και οστά και ε, σε μια πραγματικότητα και να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει από κοινού. Ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, τους σκιώδεις συζητητές και όλες τις πολιτικές ομάδες που συνεισέφεραν στην εκπόνηση της έκθεσης αυτής και στην ε, δημοτευτική αυτή εντολή όπου ελπίζουμε να έχει μεγάλη δύναμη και αποτελεσματικότητα το Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε. Και τώρα η κυρία Γεωργίευα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον κύριο Φερνάντες που παρουσίασε μια πολύ δομημένη και τεκμηριωμένη πρόταση για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις επικείμενες διαπραγματεύσεις. Όπως είπατε, πολλοί συνέβαλαν σε αυτήν την αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων που πρέπει να έχουμε, γιατί πρέπει να τις έχουμε και πώς θα αξιοποιήσουμε τις πιστώσεις που έχουμε στη διάθεσή μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υποστηρίζουμε τις προτεραιότητες που σκιαγράφησε το Κοινοβούλιο. Βεβαίως πρέπει να εστιάσουμε στην αναζωγόνηση της οικονομίας μας. Είπατε απασχόληση, επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα. Αυτά πρέπει να προωθήσουμε αν θέλουμε να υπάρξει ανάπτυξη για να έχουμε και ανταγωνιστικότητα αλλά και ευημερία. Μας στηρίξατε, στηρίξατε πολλές πρωτοβουλίες κλειδί της Κομισιόν συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος επενδύσεων. Εγκρίναμε μία τροποποιητική επιστολή που σας αποστήλαμε και χαίρομαι που βασίζεται στη συμφωνία που ε, επιτύχαμε και άρα μπορείτε να τη στηρίξετε. Και συμφωνούμε ότι πέρα από την εστίαση στην ανάπτυξη πρέπει να διατηρήσουμε την αλληλεγγύη και εντός της Ένωσης να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη και υπολογίζουν σε μας και εκτός όμως της Ένωσης. Ιδιαίτερα αυτούς που προσπαθούν να διαφύγουν από πολέμους και ιδιαίτερα όταν αυτό μετατρέπεται και εσωτερικό πρόβλημα της Ένωσης και σε εσωτερικό πρόβλημα της Ένωσης. Γι' αυτό έχουμε προτείνει τις αναγκαίες πιστώσεις πληρωμών με πολύ συγκεκριμένο τρόπο λέγοντας εδώ συγκεκριμένα πρέπει να αυξηθεί η γραμμή, ιδιαίτερα οι πληρωμές, ούτω ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες. Έχουμε 143,5 δις, 1,6% αύξηση τις πληρωμές για να μειώσουμε και τις ε, ελλείψεις πληρωμών από προηγούμενα έτη και συγκεντρωθήκαμε σε τομείς όπου οι ανάγκες είναι πιο επίγουσες και βαθιές για παράδειγμα, στο κεφάλαιο 4, 28,5% αύξηση προτείνουμε. Για τον έρασμο προτείνουμε 30% αύξηση. Και, και με βάση τη γενικότερη προσέγγισή μας, η βασική κατεύθυνση είναι να ε, εξυπηρετήσουμε τις πραγματικές ανάγκες. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και βασιζόμαστε στο Κοινοβούλιο να μας στηρίξει σε αυτήν την προσεκτική μας προσέγγιση. Και τονίζω, ότι με βάση την ενθάρρυνση του Κοινοβουλίου βελτιώνουμε τις ε, δυνατότητες προβλέψεών μας. Αυτό θα μας επιτρέψει από κοινού να κάνουμε την καλύτερη δυνατή κατανομή των περιορισμένων πόρων μας για να διαχειριστούμε τις πληρωμές στο μέλλον, ούτως ώστε να μην έχουμε αυτά που συνέβησαν το 2014. Θέλω να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να σε ευχαριστήσω για το πώς μας στηρίζετε για το διορθωτικό προϋπολογισμό και βεβαίως οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε προς τους πολίτες μας πρέπει να τηρούνται. Όταν λέμε ότι αυτό θα το κάνουμε μέχρι τότε, θα πρέπει να το κάνουμε μέχρι τότε. Όπως έχουμε συμφωνήσει και με βάση τους κοινά συμφωνημένους στόχους. Προσβλέπω λοιπόν στον επικείμενο πρώτο τριμερή διάλογος 14 Ιουλίου, εκεί από κοινού θα τονίσουμε ότι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και να μην είμαστε μόνο λόγια αλλά και πράξεις. Ευχαριστώ. Και τώρα εκπρόσωποι των διαφόρων επιτροπών του Κοινοβουλίου. Πρώτος ο κύριος Λίτς, ένα λεπτό για την Επιτροπή Ανάπτυξης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως εισηγητής της γνωμοδότησης της ΔΕΒΕΜ θέτω δύο βασικά ζητήματα. Πρώτον, οι δαπάνες για την ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να αυξηθούν κατά πολύ για το 2016 και επιγόντως η Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή είναι παγκόσμιος παράγων πρέπει να αντιμετωπίσει και τις ανθρωπιστικές κρίσεις ε, ε, η Ουκρανία, Ιράκ, Νότιο Σουδάν και Συρία. Η αύξηση λοιπόν της ανθρωπιστικής βοήθειας δεν πρέπει να γίνει μόνο στις υποχρεώσεις αλλά πρώτα απ' όλα και στις πληρωμές Μόνο έτσι μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα έχουμε τις αναγκαίες πιστώσεις αμέσως για τους ανθρώπους που έχουν βοήθεια. Δεύτερον, όλα τα κράτη-μέλη δεν τηρούν τις υποχρεώσεις του. Το 0,7% του ΑΕΠ να δίνεται για, ανθρωπιστική συνεργα... ε, συγγνώμη, για αναπτυξιακή συνεργασία. Ο στόχος αυτός έπρεπε ήδη να έχει επιτευχθεί το 2015. Η Ένωση λοιπόν πρέπει και στον προπολογισμό της να έχει αρκετούς πόρους για να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ σε ευχαριστούμε. Εκ μέρου τώρα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ε, η κυρία Κλουν, Για ένα λεπτό. Μέρος Επιτροπής έμπλε να πω ότι εμείς θέλαμε να δοθεί έμφαση ιδιαίτερα ε, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στον προπολογισμό, που είναι και μια στρατηγική την οποία ε, θέλουμε να στηρίξουμε όπως ε, και την επιχειρηματικότητα. Πώς θα τα στηρίξουμε όλα αυτά. Θέλουμε να στηρίξουμε και τις ΜΜΕ γιατί η ΜΜΕ είναι σπονδυλική στήλος και λετός των οικονομιών. Το 90% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες στην Ευρώπη. Και σε ό,τι αφορά τις μικροπιστώσεις, ε, θα στηρίξουν σίγουρα γιατί οι κυβερνήσει, οι επιτροπές, τα συμβούλια δεν δημιουργούν ε, θέσει εργασία, αλλά σίγουρα δημιουργούν ε, ένα πρόσφορο περιβάλλον ε, που μπορεί να ανθίσει εκεί η απασχόληση. Και στο τομέα τη απασχόληση έχουμε το μεγάλο, το σοβαρό πρόβλημα τη ανεργία των νέων που συνεχίσουμε να συζητούμε και θέλουμε και εκεί να υπάρξει έμφαση από την πλευρά του προπολογισμού. Θέλουμε επίση να προωθήσουμε την ανάπτυξη δεξιοτήτων ε, στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών ε, θέλουμε να αναπλάσουμε, να εξυγχρονίσουμε τα κτίρια ε, και όλα αυτά θέλουμε να περιληφθούν σε αυτή την γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριο Λαβία για ένα λεπτό εκ της τη Επιτροπή Περιβάλλοντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, σας ευχαριστούμε για όσα κάνατε αλλά νομίζω ότι ακόμα πρέπει να γίνουν πολλά και να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Φερνάντες για τη δουλειά του. Οι προπολογισμοί των τελευταίων χρόνων δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια η έλλειψη αναλήψεων πιστώσεων πληρωμών ε, δεν επιτρέπουν να ολοκληρωθούν επιτυχημένα τα προγράμματα όπως αυτό το live. Επίσης για, την, ε, για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ε, ασφάλεια των τροφίμων ε, βλέπουμε ότι τουλάχιστον θα έπρεπε να διατηρήσουμε το ίδιο επίπεδο δαπανών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ε, στο κεφαλαίο 3 για την προστασία των καταναλωτών έπρεπε τουλάχιστον εκεί να υπάρχει η απαραίτητη προσοχή ε, καθώς αυτό το κεφάλαιο αφορά την του καθημερινού βίου των πολιτών και για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς ε, η Επιτροπή ΕΜΒΗ παρακολουθεί τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς πολλές φορές λαμβάνουν και εξωτερικά κονδύλια για την εξαγωγή των δραστηριοτήτων τους. Ε, καμιά φορά όμως οι περικοπές σε αυτές τις περιπτώσεις ε, αντιτίθεται στους ίδιους τους στόχους των οργανισμών. Ευχαριστούμε και, και τώρα για την Επιτροπή Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας κυρία Φανμπόσουιτ. Σας ευχαριστώ συζητήτρια για τον ε, προϋπολογισμό 2016 στο πλαίσιο της Επιτροπής ΣΥΤΡΕ. Είμαι αντίθετο στι εξοικονομήσει που γίνονται ει βάρο του προγράμματο ερεύνη Ορίζοντα 2020 για να χρηματοδοτηθεί το σχέδιο Juncker. Πιστεύω πω αυτό το πρόγραμμα είναι ένα σαφέ παράδειγμα όπου η Ευρώπη έχει προστιθέμενη αξία. Η Φλάνδρα είναι ένα από του Ευρωπαίου πρωτοπόρου στα θέματα έρευνα και καινοτομία, κυρίω χάρη στι ευρωπαϊκέ ενισχύσει και γι' αυτό είμαι περήφανη. Θα συνεχίσω λοιπόν να ζητώ να διατηρηθεί αυτή η στήριξη. Δεν μπορώ παρά να επαναλάβω ότι είναι απαραίτητη η συνέχιση αυτών των προγραμμάτων και να επιμείνω για το ότι ε, δεν θα πρέπει να περικόπτονται τέτοια σημαντικά προγράμματα υπέρ του κοινού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Γκάλ Πέλτσε της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Ως εισηγήτρια γνωμοδότησης θα πρέπει να σας πω ότι πιστεύω πως είναι πολύ σημαντική η αγορά για και η κίνηση της αγοράς για την ε, ανάπτυξη. Είναι σημαντικό να υπάρχουν οι γραμμές του προπολογισμού για την εσωτερική αγορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάστηκε καλά και έχουμε ένα καλό πλαίσιο. Ε, σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θα ήθελα ωστόσο να διευκρινίσω ότι χρειάζεται ένας ισορροπημένος ε, προϋπολογισμός για την τελωνιακή σύνδεση και για την ε, τυποποίηση. Ωστόσο, ζούμε σε ένα περιβάλλον ε, το οποίο μεταλλάσσεται και είναι σημαντικό να επιμείνουμε για τους κανόνες ε, και είναι κάτι ακόμα που θα ήθελα να υπογραμμίσω. Οι μεταρρυθμίσεις της εσωτερικής αγοράς που φέτος ε, ε, θα γίνουν σε μεγάλο βαθμό και πιστεύουμε και ότι το φόρουμ για την εσωτερική αγορά είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ κυρία Σπυράκη της Επιτροπής Ρέτζη. Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα χρήματα που δίνονται μέσω των διαθροτικών ταμείων αποτελούν μια σημαντική, μια δραστική ενίσχυση στην οικονομική δραστηριότητα μέσω των συνεργειών στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά στην ουσία τη μοναδική πηγή χρηματοδότησης των χωρών που βρίσκονται σε κρίση και για την οικονομία και για την κοινωνική συνοχή. για να συμβεί αυτό στην πράξη επήγει να υλοποιηθεί χωρίς αποκλήσεις το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε η ευρωπαϊκή επιτροπή για τη λύση του προβλήματος με τις εκρεμείς πληρωμές από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. είναι φανερό ότι κινδυνεύουμε να βρεθούμε μπροστά σε μια χιονοστιβάδα σκεφτείτε τι συμβαίνει στη χώρα μου την ελλάδα όπου το χρηματοπιστωτικό σύστημα πάγωσε και οι πληρωμές από την ευρωπαϊκή ένωση δεν φτάνουν στους αποδέκτες. κατά την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου το 2016 οφείλουμε επίσης να λάβουμε υπόψη τα νέα δεδομένα που δημιούργησε η κρίση στις χώρες που επλήγησαν οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι το efsi θα επιστρέψει στο ακέραιο μαζί με τα κέρδη τα κεφάλαια που χρησιμοποιεί από το horizon και το ses. πρέπει να σφέψουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων φτάνουν στην πραγματική οικονομία και να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος τώρα για δύο λεπτά. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Φερνάντε που μπόρεσε να κάνει μια πραγματική διαβούλευση ανάμεσα στι επιτροπέ εν ώψη αυτού του τριμερού διαλόγου και το γεγονό ότι η Επιτροπή Προπολογισμού θα εργαστεί πάνω σε αυτέ τι γνωμοδοτήσει στι 14 Ιουλίου. Θα ήθελα να θυμίσω ποιε είναι οι προτεραιότητε σε αυτό το πλαίσιο αυτή τη διαπραγμάτευση. Καταρχήν, χρειαζόμαστε μια σταθερότητα στον προπολογισμό και ιδιαίτερα στον προπολογισμό τη Γεωργία. Είναι καλό να που δημιουργείται το, το Ταμείο ΕΦΣΥ, αλλά είναι κρίμα που για να γίνει αυτό ε, περικόπτονται άλλες γραμμές. Εγώ πιστεύω ότι αυτές θα πρέπει να προστατευτούν και κυρίως να προστατευτούν οι γραμμές της ε, γεωργίας γιατί εκεί υπάρχουν και τα αποθέματα για τις κρίσεις γιατί η γεωργία επανελειμμένες κρίσεις όπως είναι η ρωσική κρίση την οποία διανύουμε τώρα είτε θα είναι η κρίση ε, που θα προκληθεί από διάφορα από διάφορες πλευρές και πρέπει να επαγρυπνούμε και να διατηρήσουμε αυτό το αποθέμα κρίσης και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη αποθεματικά, τα ανώτατα αποθεματικά καθώς και τα προγράμματα όπως αυτό για του γάλακτος στα σχολεία. Έπειτα η Γεωργία είναι η πιο ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχουν και άλλες επί των οποίων πιστεύω θα πρέπει να προσέξουμε τα διαρθρωτικά ταμεία, ας πούμε, την εγγύηση για την νεότητα που είναι πολύ σημαντική για το μέλλον της Ένωσης και κατά αυτή, από αυτή την άποψη θα πρέπει να είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την χρηματοδότηση αυτών των αγαμών. Και τέλος το θέμα της μετανάστευσης που σίγουρα θα ξέρετε ότι εδώ και καιρό γίνεται σημαντική συζήτηση για αυτό το θέμα και πρέπει να χρηματοδοτηθεί και αυτός ο τομέας. Δηλαδή να βρεθεί μια λύση, ενώ όταν λέω να χρηματοδοτηθεί αυτό ο τομέα. Να προσέξουμε επίση ε, την έλλειψη ισορροπία ανάμεσα στι πιστώσει υποχρεώσεων και στι ε, ε, πληρωμών, στις πιστώσει πληρωμών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καντέκ δεν είναι εδώ, που ήταν η σειρά του. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής Πολιτισμού, τον κύριο Σορογεύσκη, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο πολιτισμός για τον οποίο τόσο πολύ είμαστε περήφανοι στην Ευρώπη πρέπει να τύχει υποστήριξη από όλους, όχι μόνο τα κράτη-μέλη δηλαδή, αλλά και από εμάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χωρίς ποιότητα ποιότητας, ανωτερή εκπαίδευση και συμμετοχή στο πολιτισμό δεν θα μπορέσουμε να είμαστε τόσο δημιουργικοί. Γι' αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί υπαρκή χρηματοδότηση. Στόχος μας πρέπει να είναι ένας καταναλωτής πολιτιστικών αγαθών υψηλών απαιτήσεων και κατάρτισης και καλλιέργειας που θα μπορεί να υποφελείται από το Erasmus, Erasmus Plus που έχει δημιουργηθεί για τους πολίτες της Ευρώπης αλλά φαίνεται ότι δεν του αποδίδεται τόσο μεγάλη σημασία αυτού και άλλων προ... πιλωτικών σχεδίων που δοκιμάζονται. Δεν φαίνεται να υπάρχει επαρκής υποστήριξη για πιλωτικά προγράμματα σημαντικά για τον πολιτισμό. Όπως έργα συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών για πολιτιστικές εκδηλώσεις στα πολυάριθμα φεστιβάλ που γίνονται στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους ε, των, της των Γυναικών, κυρία Ματέρα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον συνάδελφο Φερνάντες για την εργασία που κάνει και για την πεποίθηση και την αφοσίωση με την οποία ασχολείται με αυτό το θέμα. Ως εισηγήτρια της γνωμοδότησης εξ της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Δικαιωμάτων της Γυναίκας θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι αυτές θα πρέπει να προωθούνται μέσα στο πλαίσιο όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών και θα ήθελα να ζητήσω από τον συνάδελφο Φερνάντες να επιμείνει στη διάρκεια του τριμερούς ώστε να στηρίξει τα προγράμματα όπως το κόσμο που στηρίζουν την γυναική επιχειρηματικότητα και την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Και εδώ υπό το φως ε, πολλών ε, αυτοκτονιών γυναικών, ε, συγγνώμη, δολοφονιών γυναικών ή βία στην οποία υπόκειται γυναίκες θα πρέπει να στηρίξουμε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης εναντίον των στερεοτύπων σχετικά με τα δύο φύλλα και να στηρίξουμε επίσης το πρόγραμμα Δάφνη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα το λόγο παίρνουν οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων και καταρχήν ο κύριος Μπέγκε, εξ του ΕΛΚΑ, για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ρητά υποστηρίζω τον εισηγητή Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες στις προτεραιότητες που έχει ορίσει. Και θα ήθελα ιδιαίτερα να επικεντρωθώ σε αυτές που αφορούν την Επιτροπή του Εξωτερικού Εμπορίου στο κεφάλαιο 16 του προπολογισμού. Πιστεύουμε ότι ο προπολογισμό ε, πρέπει να αναγνωρίζει την ολοκεντρωμένη ε, σημασία του εξωτερικού εμπορίου και τη γεωπολιτική κατάσταση και πρέπει να έχει τη σχετική πρικοδότηση. Θεωρούμε ότι οι όλο και εντυνόμενε δραστηριότητες στον χώρο του εμπορίου, του Εθνού Εμπορίου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των Υπηρεσιών τη θα πρέπει να ε, έχουν επαρκή πρικοδότηση ώστε να μπορούν και να διαχειρίζονται τα, τις διάφορες συμφωνίες και εκ των υστέρων να αξιολογούν τη λειτουργία τους και την απόδοσή τους και να επιτρέπουν ε, την ε, τήρηση των όρων από την αξιολόγηση του ελεγκτικού συνεδρίου. Η συγκινησιακά ε, φορτισμένη συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση νομίζω απαιτεί μια επαρκή πολιτική και δημοσιότητα. Έχουμε επίσης τις ε, υπουργικές ε, διασκέψεις του κεφαλαίου 16. Έχουμε την υποστήριξη σε κράτη λιγότερο ανεπτυγμένα, τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη υποδομών και δυνατοτήτων. Η δε συζήτηση που γίνεται στο Κοινοβούλιο για την οικονομική υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλειών για την παγκοσμιοποίηση, για την διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία. Σα ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο θα λάβει ο κύριος Γκάιερ, δύο λεπτά, Σοσιαλιστέ Δημοκράτε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρία Αντιπρόεδρε, κυρία Γεωργίευα, αγαπητοί συνάδελφοι. Είχαμε στο παρελθόν πολλές αντιπαραθέσεις με το Συμβούλιο Έχω μια ισχνή ελπίδα, αλλά ελπίδα είναι πάντως ότι μπορεί να προχωρήσουμε σε μια νέα περίοδο των σχέσεών μας. Μετά την κρίση των πληρωμών, που ελπίζω να μην ξαναδούμε μπροστά μας, πιστεύω ότι μπόρεσε το Συμβούλιο να περάσει από όλες τις φάσεις της ε, ψυχοθεραπείας, από το διαφωτισμό, την κάθαρση, την αρχή της ε, ίασης. Ελπίζω ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια κατάσταση όπου μέσα σε λίγες εβδομάδες μπορούν να προχωρήσουν σε μια επισκόπηση του πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η κρίση πληρωμών τα θεσμικά όργανα και η Λουξεμβουριανή Προεδρία, αγαπητοί συνάδελφοι, ελπίζω ότι μπορεί να υπενθυμίσει τι έχει και να θυμηθεί τι έχει ε, συμφωνηθεί η πολετονική Προεδρία. Όταν δηλαδή πάει να κοιτάξει τα θέματα αυτά για άλλη μια φορά το Συμβούλιο, θα τα κοιτάει πάλι αφαίρετα όπως είχαμε και στο παρελθόν διαπιστώσει ή θα ε, τηρήσει μία γραμμή προτεραιοτήτων αναγνωρίσιμη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αγαπητοί φίλοι. Δεν με εκπλήσει το γεγονό ότι η πρόταση του προπολογισμού που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απόκληση 10 δισεκατομμυρίων ανάμεσα στι δεσμεύσει υποχρεώσεων και τι πληρωμέ, στι αναλήψει υποχρεώσεων και τι πληρωμέ. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίε και κύριοι, έχει να αντιμετωπίσει όλο και μεγαλύτερε δυσκολίες. Τις συζητάμε σε κάθε σύνοδο μέλη του Κοινοβουλίου και μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή, μετά το failing state, τη Λιβύη, την, την Ουκρανία και άλλα αντίστοιχα προβλήματα που δεν χρειάζεται να σα αναφέρω διεξοδικά. Βλέπουμε ότι η εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει αποτελεσματικά μέσα. Αυτό δεν θα εξαρτηθεί μόνο από τα χρήματα, αλλά χρειάζονται και τα χρήματα και αυτό ισχύει και για τα μέσα που θα αναπτύξουμε για τη μεταναστευτική πολιτική. Έχουμε μια επιπλέον πρόκληση τώρα όμως. Το ΕΦΣΙ, το πρόγραμμα Juncker που πρέπει να ενσωματωθεί σε αυτόν τον προϋπολογισμό που σημαίνει ένα δισεκατομμύριο ακόμη ε, από το ε, αποθεματικό και πέντε δισεκατομμύρια από τον τρέχοντα προϋπολογισμό πρέπει να αντληθούν και να χρηματοδοτηθεί αυτό το πρόγραμμα επενδύσεων. Ε, πρέπει λοιπόν να μιλούμε για χρήματα βεβαίω, αλλά και για την πολιτική εικόνα και διαμόρφωση του προπολογισμού και έτσι μπορούμε να περάσουμε σε μια νέα φάση. Ευχαριστώ πολύ. Μέλ, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ την Αντιπρόεδρο Γεωργιέβα για την ε, εξαίρετη συνεργασία κατά την εκπόνηση της, της προτάσεως. Εμείς ως ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών βλέπουμε ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε καλά βήματα προόδου προς την ορθή κατεύθυνση με τον προϋπολογισμό αυτό. Ταυτόχρονα όμως μας λυπεί το γεγονός ότι εν τέλει παραμένει το status quo ιδιαίτερα και με όλη την εκτίμηση θα πρέπει να φέρω αντίλογο στον αγαπητό συνάδελφο κύριο Γκάιερ ως προς την ιατρική του ανάλυση. Δεν βλέπω δηλαδή πράγματι το πρόβλημα των ε, μη εξοφληθισών ε, πιστώσεων, των μη ε, εξοφληθισών υποχρεώσεων να έχει επιληθεί με τα 143 δισεκατομμύρια, γιατί μας λείπουν 110 δισεκατομμύρια, τα οποία δεν μπορούμε να τα βρούμε από το πουθενά. Πολύ θα χαιρόμουν λοιπόν, εάν είχαμε στο Κοινοβούλιο το θάρρος να προχωρήσουμε σε μια μεταρρύθμιση που δεν θα σήμαινε μόνο άθροισμα πολλών λογαριασμών και εν τέλει εξόφληση όποιου μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ. Αλλή δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή, του κύριο Φερνάνδε. Είναι μια πολύ συγκροτημένη έκθεση, αλλά να σας πω πως στην 16η ε, αναθεώρηση αυτό στο οποίο καταλήξαμε είναι ότι ναι, συνάδει και η ανάληψη υποχρέωσεων έχει μειωθεί 5,2%, οι πραγματικές πληρωμές αυξάνονται 1,1%. Άρα λοιπόν έτσι θα μειώσουμε τις καθυστερήσεις και θα είμαστε βιώσιμοι μέχρι το 2016. Άρα λοιπόν ε, ε, ιδιαίτερα εκτιμήθηκε η συνεργασία μεταξύ της Σχετικής Επιτροπής και της Επιτρόπου Γεωργίευα έτσι ώστε ε, να προχωρήσουμε από το στομείο στο οποίο βρισκόμαστε στην αρχή της θητείας. Έχουμε την ψηφιακή ενιαία αγορά, τις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αύξηση ανταγωνιστικότητα της στήριξης στους γεωργούς, όπως επίσης και τις ε, πληρωμές προς το επενδυτικό ταμείο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης, γιατί μέσω αυτού του προϋπολογισμού θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την πρόκληση της μετανάστευσης. Όμως οι μεταναστευτικές ώρες αυξάνονται συνέχεια και ίσως τα όρια που έχουμε θέσει να έχουν ήδη ξεπεραστεί. Και επίσης θα πρέπει να πούμε πως οι καθυστερήσεις που έχουμε ήδη συσσωρεύσει μαζί και με τον πληθωρισμό ε, που αυξάνεται ε, οδηγεί στο συμπέρασμα πως πραγματικέ αυξήσεις δεν θα έχουμε. Άρα λοιπόν ο προπολογισμός μένει περίπου στα επίπεδα που ήταν. Είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή για να μειώσουμε κατά 4% τους πόρους για την κοινωνική συνοχή όταν αυτή τη στιγμή αυξάνονται οι διαφορές μεταξύ περιφερειών και κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κοινικέ γραμμές στηρίζουμε τις βασικές γραμμές του προπολογισμού καινοτομία, θέση εργασία ανταπόκριση στις προκλήσεις μετανάστευσης, όπως επίσης και ανάπτυξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σίγουρα θα έχουμε το πιο θετικό αποτέλεσμα μετά από την όλη διαδικασία του τριμερούς διαλόγου. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νίριάντα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Φερνάντες για τη σκληρή δουλειά που έκανε στην έκθεση αυτή και νομίζω ότι πολλά από τα σημεία τα οποία έχει συμπεριλάβει θα μας βρούνε σύμφωνους. Πρέπει να σου πω βέβαια πως η εντολή για το 2016 έχει βελτιωθεί. Δεν έχουμε όμως μεγάλες διαφορές, λιτότητα, αρνητικές πολιτικές και μια νεοφιλελεύθερη προσέγγιση ε, που προωθείται. Η πρόσφατη κρίση στην Ελλάδα δείχνει πως θα πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτό το εσφαλμένο μονοπάτι και θα πρέπει να προσφέρουμε ε, και θέσεις υψηλής ε, ε, ποιότητας στον εργασιακό χώρο αλλά και ευφύ ανάπτυξη πολιτικής συνοχής. Ένας φάκελος πολύ σημαντικός. Θα πρέπει να στηρίξουμε τις χώρες οι οποίες αγωνίζονται γιατί αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους περιορισμούς. Ξέρετε, ε, μετά από τα προβλήματα που είχαμε με το δημοσιονομικό πλαίσιο του 2013 μας κούρασαν και είπαμε πως το επόμενο θεματολόγιο ε, θα πρέπει ε, να κάνουμε μια μεγαλύτερη προσπάθεια, μια αναθεώρηση έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στα όσα περιμένουν από εμά οι πολίτες. Ο κύριος Μαραγκάλ είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Το καλύτερο που θα μπορούσε να δηλώσει κανείς για αυτό τον προϋπολογισμό, κύριε Φερνάντης, κυρία Γεωργίεβα, είναι πως τουλάχιστον δεν θα είναι ιδιαίτερα βλαβερός για κανέναν. Είναι ορθός, ισορροπημένος, ε, προσφέρει τα κατάλληλα εχέγγυα και εμείς μέχρι την τελευταία στιγμή θα αγωνιστούμε όπως κάθε φορά και θα καταλήξουμε σε μια τίμια συμφωνία. Τώρα αυτό το 1,6 και το 4% που είναι τα αντίστοιχα στην ανάληψη υποχρεώσεων και πληρωμές δεν μπορώ να σας πω πώς σημαίνουν πραγματικά ε, κάποια αύξηση. Έχουμε μια σημαντική περικοπή των ε, πληρωμών ε, γιατί έχουμε αυτές τις καθυστερήσεις και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια με τα προγράμματα του 2014 και 2020 όταν όλα τα προγράμματα αρχίσουν να εφαρμόζονται. Πρέπει να σας πω πως έχουμε το θέμα του πρασινίσματος, του greening του προϋπολογισμού και αυτό είναι καλοδεχούμενο, αλλά αν αφήσουμε αυτό το θετικό να δούμε ποιο είναι το αρνητικό στοιχείο, ε, στηρίζουμε το ITER, το πρόγραμμα αυτό. 500 και εκατομμύρια για ένα ε, ε, πρόγραμμα που είναι πιο ανισχυτικό και πιο αμφισβητήσιμο παρά θετικό. Τώρα, για τα 2013 και τις καθυστερημένες πληρωμές, ας τελειώσουμε με αυτό και συζητήσουμε τα υπόλοιπα. Τώρα έχουμε και ένα άλλο θέμα, πολύ πιο σημαντικό, γιατί ξέρετε, όπως και η ορχέστρα του Τιτανικού, εμείς συνεχίζουμε με τα τραγούδια μας, με τη μουσική μας και γύρω-γύρω υψώνονται φωνές που ζητούν άλλες αποκρίσεις από εμείς, πιο φιλόδοξες, πιο ουσιαστικές. Η συζήτηση για την ε, Ελλάδα που έγινε σήμερα εδώ αποδεικνύουν πως πραγματικά αντιμετωπίζουμε αντιφάσεις. Οι ΙΠΑ έχουν ένα προϋπολογισμό που είναι γύρω στο 20% του ΑΕΠ και εμείς είμαστε ακόμα στο γύρω στο 1% του ΑΕΠ της Ευρώπης. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Είναι καλός και ορθός ο προϋπολογισμός, αλλά δεν δίνει ε, τα εργαλεία που χρειάζεται η Ευρώπη για να αναπτυχθεί οικονομικά και να αντιμετωπίσει τις ανισότητες που βρίσκουμε σήμερα μας. Ο κύριος Άρνοτ είναι ο επόμενος ομιλητής, λέει ο πρόεδρος. Όταν έχεις ε, χαράξει ρότα για το παγόβουνο, δεν θα έπρεπε ο καπετάνιος να λέει «ακολουθήστε τα όσα βλέπετε στο χάρτη». Νομίζω ότι ε, εδώ κάνουμε κάποιες ταχυδακτηλουργίες, γιατί βλέπουμε τι γίνεται με την αύξηση του ΑΕΠ, βλέπουμε ποια είναι τα φερολογικά μας έσοδα, βλέπουμε ποιο είναι το κόστος της συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στις χώρες μας ένας ίδιος προϋπολογισμός για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που παραμένει ίδια. Τι μας διδάσκει το ελληνικό θέμα. Πως δεν μπορούμε να συνεχίζουμε ακολουθώντας τις παλιές μας τακτικές. Έχουμε εδώ την Ευρωπαϊκή Αρχή της όλο και πιο στενής ένωσης. Βλέπετε κάτι τέτοιο εδώ, πετυχαίνουμε κάτι τέτοιο. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο αποτελεσματικά. Νομίζω ότι οποιοδήποτε κράτος θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα σε επιδόσεις από ότι η γραφειοκρατία των Βρυξελών, αν κρίνουμε από τα αποτελέσματα. Ε, ο κύριος, κυρία Μοντέλ για ένα λεπτό. Το σχέδιο προπολογισμού 2016 αντικατοπτρίζει τη θέση α, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει κάντε αυτό που λέω, όχι αυτό που κάνω. Έχουμε μείωση 2,2% στην, στην Κομισιόν και 2,4% για το Κοινοβούλιο. Η Κομισιόν θα έπρεπε να αυξήσει του, ε, τους μισθούς του προσωπικού κατά 5,4%. Οι Βρυξέλλες θα έπρεπε να επιβάλλουν τη λιτότητα στον εαυτό τους πριν την επιβάλλουν σε άλλους. Γιατί μεταξύ, ε, μειώνεται η εσωτερική ζήτηση στα κράτη-μέλη και με το σχέδιο Juncker που αναμένεται ως μεσίας από τους θειασότες του Ευρωπαϊκού Νηπιαγωγείου δεν ε, πρόκειται να καταφέρει να κάνει κάτι καλύτερο. Εν τω μεταξύ προβλέπουμε βοήθεια χρηματική για την Ουκρανία που είναι εκτός από Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά αρνούμεθα τη βοήθεια ε, στην Ελλάδα. Τελευταίο αστιάκι, ε, έχουμε και μιλάμε για, για δικαιώματα του ανθρώπου, ενώ ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Σούλτς μιλούσε για τέλος εποχή ΣΥΡΙΖΑ και ήταν έτοιμος να αντικαταστήσει την κυβέρνηση. Ευχαριστώ κύριο Σπρέντα για, δύο, ε, για 1,5 λεπτό. Να, συγχαρώ τον κύριο Φερνάντες που συνέταξε την ε, έκθεση που έλαβε υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των διαφόρων επιτροπών και να εκφράσω την ικανοποίησή μου όσον αφορά την σημαντική αύξηση στο σχέδιο της Επιτροπής για τις πιστώσεις πληρωμών και πιστώσεις υποχρεώσεων για την εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Είμαι πεπισμένο ότι για να μπορέσει η Ένωση να έχει ε, τη θέση που τη αναλογεί παγκοσμίω θα πρέπει να έχει και τα μέσα που χρειάζονται γι' αυτό. Και γι' αυτό και οι προστιθέμενοι πόροι που προβλέπονται στον προπολογισμό από την Κομισιόν θα πρέπει να διατηρηθούν στο τελικό ε, προπολογισμό. Να διατηρηθούν αυτέ οι αυξήσει είναι πολύ σημαντικό για τι πιστώσει πληρωμών, γιατί σε αντίθετη περίπτωση μια ολόκληρη σειρά προγραμμάτων τη Ένωση, όπω το Μέσο για τη Σταθερότητα και την Ειρήνη, θα έχουν ε, δυσκολίε να επαναλάβουν ε, τι δραστηριότητέ του που εν μέρει έχουν διακοπεί για λόγω οικονομικών δυσκολιών. Στην εξωτερική πολιτική το κοινοβούλιο μας ε, θα συνεχίσει να είναι δεσμευμένο και προσιλωμένο στην ανάπτυξη των γειτονικών σχέσεων προς τα Νότο και προς τα Ανατολάς για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις χώρες που μας περιβάλλουν. Θεωρώ επίσης ότι είναι σημαντικό ο φετινός προπολογισμό να δείξει τη δέσμευσή μας στην σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις χώρες γύρω μας, αλλά και πιο πέρα, πιο μακριά και ο προπολογισμό μας θα πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτούς τους ε, ε, προβληματισμού που βρίσκονται στο επίκεντρο ε, των ανησυχιών μας. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Τόμας, δύο λεπτά. You have to... Uh, okay. Okay. She will come afterwards. Καλώς, θα έρθει τώρα Ashworth. Δύο Η έκθεση αναφέρεται στη λογοδοσία, την αξιοποίηση των πόρων, μεγάλα για τα μεγάλα, μικρά για τα μικρά. Πολύ ενθαρρυντικά όλα αυτά. Και γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτρόπο Τζορτζίεβα, η οποία εισάγει τι έννοιε τη κοινή λογική και τη πειθαρχία στη διαδικασία του προπολογισμού. Έχω όμω μια ανησυχία. Το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για τις λεπτομέρειες της διατύπωσης του προϋπολογισμού. Αλλά πολύ λίγο ενδιαφέρεται για τις επιδόσεις και την απόδοση του προϋπολογισμού. Αυτό δεν είναι παραδεκτό. Οι οποίοι συνάδελφοι δαπανούνται, δαπανούνται χρήματα του Ευρωπαίου φορολογουμένου. Αλλά δεν κοιτάμε να δούμε αν δαπανήθηκαν όσα έπρεπε, ούτε όπως έπρεπε, ούτε εκεί που έπρεπε. Και γι' αυτό πολύ συχνά οι αποφάσεις μας στηρίζονται σε πολιτικές παραδόσεις και πολύ σπάνια σε αποδεικτικά στοιχεία και ουσία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δεπρέ για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα σας εξπλήξω αν πω ότι θέλω να υποστηρίξω πλήρω τον συναδελφό Ζωζέ Φερνάντε στην έκθεση του για τον προπολογισμό και ιδιαίτερα θέλω να τονίσω τη σοβαρότατη και πολύ καθαρή προτεραιότητα που δίνει στην ανάπτυξη, την απασχόληση που χρειάζονται η Ευρώπη. Η Ευρώπη χρειάζεται την ε, ανάπτυξη όσο χρειάζεται άνθρωπο στο ψωμί και γι' αυτό θα έλεγα ότι πρέπει να έχουμε την τροφοδότηση των ε, ταμείων που είναι σχετικά με τις στρατηγικές επιλογές, όπως επίσης πρέπει να διατηρηθεί και ο ορίζον 2020 και η συνδεσιμότητα στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα επίσης θέλω να υποστηρίξω την ε, δέσμευση των ποσών για τη μεταναστευτική πολιτική και ιδιαίτερα την ισότιμη κατανομή μεταναστών και ετούντων το άσυλο καλύτερα στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι βρίσκω σκανδαλώδο το γεγονό ότι ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία ε, λέμαργα βάζουν στην τσέπη τα διαρθρωτικά κονδύλια αρνούνται να δεχθούν μερικές δεκάδες έστω ετούντων το άσυλο στην επικρατεία τους για να του φιλοξενήσουν. Επίσης θα συμφώνησα με τον εισηγητή ότι χρειάζεται να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια, όπω πρότεινα ε, πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η τρομοκρατική απειλή είναι πραγματική απειλή και θα παραμείνει η υπαρκτή απειλή. Χρειάζεται λοιπόν να ενισχυθούν ε, οι κατάλληλε αρχέ και φορεί και ιδιαίτερα η Europol με τα μέσα που απαιτείται. Και απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να τεθεί εν τέλει τέρμα στο ηλίθιο που θα, όπως θα το ονομάζω σύστημα τον έχουν οι, προτερ... οι υπηρεσίες οι αποκεντρωμένες ε, την πλήρη απαλλαγή από τον προτερισμό προτεραιοτήτων και λογοδοσίας. Ευχαριστώ πολύ Ορμπάν. Κύριε Φερνάντες. Εμάς, η δική μας ομάδα παρουσίασε πάρα πολλές τροπολογίες. Κάποιες έχουν γίνει αποδεκτές και κατά τη γνώμη μου βελτιώνουν το κείμενο. Παρ' αυτά θα επαναλάβουμε στην γενικότερη κριτική που ασκούμε σε αυτό το σχέδιο προπολογισμού πως είναι υπερβολικά αυστηρός και ανεπαρκής και δεν ανταποκρίνεται στο ύψος των προκλήσεων που δημιουργεί η κρίση που αντιμετωπίζουμε και που εμβαθύνεται από τις περικοπές και από την πολιτική λιτότητα Χωρίς φιλοδοξία, χωρίς δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας ποιοτικέ και εάν δεν αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο που να μην βασιζόμαστε πια σε ορεικτά καύσιμα, θα έχουμε προβλήματα στην Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τότε τα πραγματικά κοινωνικά δράματα που θα βιώνει καθημερινά ο πληθυσμό μας. Ο ελληνικός λαός είπε απερίφραστα πως φτάνει πια στην πολιτική αυτή και στην Ευρώπη της λιτότητας. Εσείς έχετε την υποχρέωση να τους ακούσετε, να ακούσετε τους λαούς της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χούμπνερ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Εκ μέρους της Επιτροπής ΑΦΚΟ ε, πρέπει να σας πω πως εμείς δεν είμαστε ε, ιδιαίτερα, δεν εμπλεκόμαστε ιδιαίτερα στο θέμα αυτών των προϋπολογισμών, αλλά για την Επιτροπή ΑΦΚΟ πρέπει να σας πω έχουμε το πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους πολίτες», «Europe for Citizens», για το οποίο η Επιτροπή έχει αυξήσει τη χρηματοδότηση και ελπίζουμε πως αυτή η χρηματοδότηση δεν θα περικοπεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ζούμε σε δύσκολες συνθήκες, υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης. Πρέπει εμείς να στραφούμε προς τους πολίτες, να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη και να βελτιώσουμε την αλληλοκατανόηση. Και μέσω αυτού του πρόγραμμα μπορούμε να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία. Δεύτερον, έχουμε τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών. Ένα ουσιαστικό ε, εργαλείο για την συμμετοχική δημοκρατία. Αυτή η πρωτοβουλία λοιπόν θα πρέπει να γίνει πιο ορατή στον προπολογισμό. Εκεί προτείνουμε να δημιουργήσουμε μία υπογραμμή η οποία θα είναι ε, δημοσιονομικά ουδέτερη αλλά θα μας επιτρέψει να έχουμε μεγαλύτερη ορατότητα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μούντι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φερνάντες για όλη την προσπάθεια που έχει κάνει για την εντολή αυτή και να καλωσορίσω την προσέγγιση της, κυρίας, της Επιτρόπου κυρίας Γεωργίευα που θέλει να αναθερμάνει την οικονομία. Αλλά δεν θα πρέπει απλώς να παρακολουθούμε τι γίνεται σήμερα στην οικονομία. Θα πρέπει να διαμορφώσουμε την οικονομία του μέλλοντος. Και για το λόγο αυτό το προπολογισμό για το Horizon 2020 είναι τόσο σημαντικός και θα πρέπει ο τριμερής διάλογος για τον προπολογισμό του 2016 να ενισχύσει το κομμάτι αυτό. Έρευνα, και καινοτομία στηρίζονται από το Horizon 2020 και αυτά είναι τα μέσα μέσω των οποίων μπορούμε να εξασφαλίσουμε ποιοτικέ θέσει εργασία για το μέλλον. Ένα μέλλον το οποίο ε, θα φέρει τεράστια τεχνολογική αλλαγή και μέσω αυτού του κλάδου μπορούμε να πετύχουμε οι γενιές που θα μας ακολουθήσουν να έχουν τις θέσεις εργασίας που τους είναι τόσο απαραίτητες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κοσμιούκ για ένα λεπτό. Ο κύριος Κοσμιούκ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Επίτροπε, θα ήθελα να τονίσω ότι οι πιστώσεις υποχρεώσεων 153 εκατομμυρίων ευρώ ενώ οι πιστώσεις πληρωμών 10 εκατομμύρια λιγότερα αν το συγκρίνουμε με το 2015. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρόκειται για 2,4% διαφορά που ουσιαστικά δείχνει ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη. Η Κομισιόν λοιπόν ίσως δυσκολευτεί να κάνει όλες τις πληρωμές ενώ στον τριμερή ακούσαμε ότι οι πληρωμές θα μειωθούν από 24 κατά 24 δις το 2014 και 2 δις το 2015, δηλαδή μεγάλη μείωση που είναι επιθυμητή, ωστόσο χωρίς υψηλή αναλογία των πιστώσεων πληρωμών θα έχουμε πρόβλημα, διότι όλες αυτές οι εκκρεμείς πληρωμές αφορούν τις προηγούμενες προοπτικές. Θα έχουμε τεράστιες καθυστερήσεις δηλαδή στη χρηματοδότηση. Ο κύριος Όλμπριχτ. Πρόεδρε, Επίτροπε. Το 2016 θα είναι εξαιρετικά σημαντικό έτος από την άποψη του προϋπολογισμού. Καταρχήν, θα πρέπει να ελέγξουμε αν οι θεσμικές μας συμφωνίες λειτουργούν καλά όσον αφορά τις πληρωμές γιατί το 2016 οι εκκρεμείς ε, ε, πιστώσεις πληρωμών θα πρέπει να μειωθούν στα 2 δις και θα πρέπει να, βρούμε, να δούμε πώς θα λειτουργήσει ο νέος τρόπος εργασίας που έχει εισαχθεί. Μόνο το 2016 δε θα δούμε το, τις πρώτες επιπτώσεις του Ταμείου Γιούνκερ, του σχεδίου Γιούνκερ όπως λέγεται το 2016. Επίσης θα έχουμε και τις πρώτες επιπτώσεις από των ε, δημοσιονομικές προοπτικές 2014 με 2020, το νέο πλαίσιο δηλαδή, και ελπίζω ότι θα δούμε και τις πρώτες πληρωμές, διότι... Ε, δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν τόσο πολλά ράλς όπως παλιότερα. Πρέπει λοιπόν να αναζωογονηθεί και να αλλάξει ο προπολογισμό μα. Τώρα το πώ θα χαρακτηριστούν τα χρήματα του προπολογισμού του 2016, πολλά θα εξαρτηθούν από το όραμα που θα δώσουμε. Ευχαριστώ. Νεγκρέσκου. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Προσέρχεται στον τριμερή διάλογο με ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Είναι πολύ σημαντικό για μας η δημοσιονομική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι αρθρωμένη ε, πάνω στις ε, επενδύσεις, πάνω στο μέλλον για να εξασφαλίσουμε το μέλλον των πολιτών. Χρειάζεται ένας προϋπολογισμό λοιπόν ο οποίος θα ξεφεύγει από την πολιτική και τη λογική της ε, λιτότητας και που θα εξασφαλίζει επενδύσεις για τους ανθρώπους, για να δημιουργούνται θέσεις εργασίας, για να υποστηρίζεται η επαγγελματική κατάρτιση, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ανάπτυξη της δημοκρατίας στην Ευρώπη και ο ενεργός ρόλος μας ε, στην προαγωγή των αξιών μας. Γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πιο σαφή αποτελεσματικά και ξεκάθαρα τις ε, δαπάνες ε, του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και με τη λύπη που έχω να εκφράσω για την απουσία των εκπροσωπών του Συμβουλίου για άλλη μια φορά σήμερα από εδώ ε, θα πρέπει και το Συμβούλιο να ακολουθήσει τις αρχές. Ευχαριστώ πολύ. Μαρινέσκου, ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε. θα διαπραγματευτείτε με τον κύριο Φερνάντε στο πλευρό σας στον προπολογισμό του 2016. Τον γνωρίζετε καλά τον κύριο Φερνάνδε. Είχατε την ευκαιρία να διαπραγματευτείτε μαζί του το Ταμείο Επενδύσεων, των Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΥ. Και θεωρώ ότι ο προπολογισμό του 2016 θα είναι ε, σημείο αναφορά. Γιατί θα είναι η πρώτη φορά που θα ενσωματωθούν πληρωμές στα διευθυντικά ταμεία και επίσης θα πρέπει να καλύψουμε τα 25 δισεκατομμύρια των ενεξόφλητων λογαριασμών από το Ταμείο Συνοχής και να αντλήσουμε τα κονδύλια για τον ορίζοντα 2020 και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θα έχουμε λοιπόν μια πολύ περίπλοκη κατάσταση. Θα έχετε μια πολύ περίπλοκη κατάσταση να αντιμετωπίσετε. Είδατε ποια είναι η θέση του εισηγητή μας. Είναι στέρεα εδρεωμένη. Έχει περιγράψει πολύ σωστά τον προπολογισμό και τις διαπραγματεύσεις του και ελπίζω ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν θα ακολουθήσουν την πεπατημένη. Δηλαδή τελευταίο, το τελευταίο βράδυ το Συμβούλιο να λέει όσο εδώ και με παρέκει και να υποχρεούνται οι πάντες να τον δεχθούν τον προπολογισμό αυτό ή δάλλως δεν θα έχουμε προπολογισμό για την επόμενη χρονιά. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία στον προπολογισμό, δηλαδή και να εξοφληθούν οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί και να υπάρξουν πληρωμές για την πολιτική συνοχή για το 2020 και, το 2020 και να αντιληθούν τα κονδύλια για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και πρέπει ασφαλώς να παραδεχθούμε την πραγματικότητα στην πραγματικότητα, εάν έρθει η ώρα, ότι δεν θα έχουμε προπολογισμό 2006 αν δεν ληφθούν οι κατάλληλε αποφάσει. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Η κυρία Τωμά δεν είναι ακόμα στην Α, όχι, εδώ είσαστε. Καλώ την. Ε, πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ, κυρία Επίτροπε. Ζητώντα συγγνώμη, γιατί αυτή η μέρα έχει πολλέ ιδιαιτερότητε και δυσκολίε για μένα. σω, ε, κυρία Επίτροπε, θεωρήσετε ότι είμαι κακόπιστη. Η... Καθυστέρηση όμω. Στην υλοποίηση των ε, προγραμμάτων με συγχρηματοδότηση έρχεται ακριβώς στη στιγμή που χρειάζεται για να καλύψουμε τους ανεξόφλητους λογαριασμούς μας. Ε, προτείνει μια ριζική μείωση μέχρι τα 2 δισεκατομμύρια η Επιτροπή για τους ανεξόφλητους λογαριασμούς. Πολύ ωραία. Αλλά τα κράτη-μέλη τι θα κάνουν, θα συμφωνήσει τελικά το Συμβούλιο να εξοφλήσει αυτού του λογαριασμού, αυτά τα χρέη. Γιατί βλέπουμε χρόνο το χρόνο η έννοια τη ευθύνη ε, του Πάκτα Sunt Servanda, τη υπευθυνότητα τελευταία ανάλυση, να μην είναι προτεραιότητα για τα κράτη και τι κυβερνήσει του. Επίση έχουμε τα 10 δισεκατομμύρια απόκληση ανάμεσα σε αναλήψει υποχρεώσεων και τι πληρωμές. Κακό ιονός για το σχέδιο για την ε, αντιμετώπιση της κρίσης πληρωμών δεν ήταν ένα ε, εφεύρημα, ήταν μια πραγματικότητα. Και τώρα έχουμε και ένα άλλο μέσο που έχουν ανακαλύψει τα κράτη-μέλη, μέχρι τα τελευταία στιγμή δηλαδή να μην εξοφλούν του λογαριασμού, ένα τρόπο ε, που έχουν ανακαλύψει για να κάνουν οικονομίε από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Το πολιετέ ε, δημοσιονομικό πλαίσιο έχει ξεπεραστεί. Το ίδιο και ο προπολογισμό με τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνεται. Γνωρίζουμε ποια είναι τα όρια το εγχειρήματο, γιατί μπορεί να είναι αυξημένη η πρικοδότηση του υπολογισμού αλλά παραμένουν τα 2 δισεκατομμύρια του παθηματικού, σαν να μην χρειαζόταν επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο υπολογισμό δίνει τις, ε, την έμφαση στι ε, δράσει προτεραιότητα. Πολύ καλά, αλλά χρειάζονται οι πραγματικέ ανάγκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να ικανοποιηθούν και δεν προβλέπεται ούτε μία δεκάρα ούτε ένα λεπτό του ευρώ για να βοηθήσουμε τα 5 εκατομμύρια ε, νέων που βρίσκονται σε απόγνωση. Μια φράση ακόμα λέει ο πρόεδρος, καλώς τελειώσω. Σας ευχαριστώ θερμά. Και τώρα ο κύριος και ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην ε, κυρία Επίτροπο γιατί Δημιούργησε το κατάλληλο περιβάλλον για να γίνουν διαπραγματεύσει και να συνεργαστούμε μεταξύ μα. Την ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερα που τόσο τακτικά έρχεται στο Κοινοβούλιο για να συζητήσει τα θέματα αυτά μαζί μα. Επίση θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φερνάντε, τον εισηγητή, γιατί ήρθε στη συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, εκεί εγώ είμαι εισηγητή για το θέμα αυτό και θα ήθελα τέλος μετά τις ευχαριστίες να σχολιάσω και το θέμα του προπολογισμού. Το να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας είναι ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το λόγο αυτό πιστεύω πως ε, τούτος εδώ ο προϋπολογισμός δεν θα πρέπει να υποχρηματοδοτείται με τον ίδιο τρόπο που σημαίνει σήμερα. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αυξήσει τους ε, πόρους που υπάρχουν για σημαντικές ε, υπηρεσίες όπως η Frontex, η Europol και είναι προφανές πως ε, υπάρχει μια έλλειψη πόρων η οποία θα συνεχιστεί. Είναι απαράδεκτο ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να διαθέτει μόνο το 1% για θέματα ασφάλειας. Θα πρέπει να προβληματιστούμε για το πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια όταν είναι τόσο χαμηλή η πόρη, γιατί χωρίς την κατάλληλη χρηματοδότηση δεν είναι ε, δυνατόν κάτι τέτοιο. Ελπίζω πως στην διαπραγματευτική εντολή αυτό θα ε, ληφθεί υπόψη. Βάντε Κάμπ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας πω πως η εμπιστοσύνη μου στο πρόσωπο του κυρίου Φερνάντες είναι τεράστια και εξίσου πιστεύομαι και την κυρία Γεωργίευα. και νομίζω ότι μπορείτε να οδηγήσετε αυτό το φάκελο σε ασφαλές λιμάνι. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο. Το Συμβούλιο ζητά από την Ευρώπη να κάνει όλο ένα και περισσότερα αφενός. Αλλά όταν καλείται να πληρώσει το λογαριασμό εμφανίζεται ιδιαίτερα διστακτικό αφετέρου. Εμείς θα μπορούσαμε να γίνουμε πιο αξιόπιστοι. Εάν χρειάζεται να αναλάβουμε νέα δράση, τότε θα πρέπει να αφήσουμε πίσω κάποιες δράσεις ε, και να το κάνουμε αυτό με μεγαλύτερη αυστηρότητα. Δηλαδή, αιτήσεις δαπάνης είναι πάντα χαμηλότερες από αυτές που έχουν προϋπολογιστεί. Για την περσινή χρονιά, να σας πω, πως θα μπορούσαμε αυτά τα κονδύλια να τα είχαμε χρησιμοποιήσει για να καλύψουμε καθυστερήσεις ε, στις πληρωμές και να μην επιστρέψουμε τα χρήματα αυτά στα κράτη-μέλη. Έχουμε κάποιο περιθώριο στον προϋπολογισμό και θα πρέπει το δημοσιονομικό πλαίσιο να γίνει πιο ευέλικτο. Εγώ εδώ προσωπώ το ΕΛ και για θέματα μεταφορών και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η σχέση μεταξύ της διευκόλυνσης και του νέου πακέτου, του μηχανισμού δηλαδή και ε, του καινούριου πακέτου. Γιούνκερ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Καντέκ, για ένα λεπτό. Ο κύριος Καντέκ, με συγχωρείτε, σας ευχαριστώ όλους για την πολύ καλή δουλειά που κάνατε και βλέπω πως ε, η εντολή και το σχέδιο εντολής είναι αρκετά κοντά σε αυτά τα οποία είχαμε πει εμείς για θέματα γεωργίας και κυρίως αλίας, δηλαδή εξυγχρονισμός του στόλου, προσπάθειες που γίνεται για την αλφιετική δυνατότητα και δυναμικότητα είναι πολύ σημαντικά θέματα. Αλλά όπως ξέρετε και εσείς, για την Επιτροπή Αλίας είναι πολύ σημαντικό αυτά τα κονδύλια να επιτρέπουν να εφαρμόσουμε στην πράξη την κοινή αληθική, πολιτική. Και βλέπετε πως έχουμε ε, πως έχουμε ε, κονδύλια τα οποία διατίθενται για διεθνή συμφωνία τα οποία δεν έχουν αυξηθεί καθόλου. Και πώς θα πετύχουμε τους στόχους της αναθεώρησης τότε δηλαδή για την βιώσιμη απόδοση και τα όσα έχουμε θέσει για το 2015. Πώς θα συλλέγουμε δεδομένα, πώς θα ελέγχουμε την αλία έτσι ώστε να γίνουν σεβαστοί και να εφαρμοστούν σωστά οι κανόνες της πολιτικής αλίας. Περιμένω να δω τι θα πει το Συμβούλιο γιατί δεν θέλω να έχουμε καμία μείωση σε σχέση με την πρόταση της Επιτρόπου κυρία Γεωργίευα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακολουθήσουμε τώρα τη διαδικασία Catch the Eye. Έχουμε αρκετούς συναδέλφους οι οποίοι έχουν εγγραφεί. Ο κύριος Νοβάκοφ είναι ο πρώτος ο οποίος θα μιλήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Όσοι βρίσκονται εκτός αυτής της αίθουσα, πολύ συχνά δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τα στοιχεία και τα δεδομένα που παρουσιάζουμε. Τους ενδιαφέρουν μόνο τα αποτελέσματα. Και νομίζω ότι αυτός είναι από τους πρώτους πολυπολογισμού που βασίζονται σε αποτελέσματα. Αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις. Κατάσταση στην Ελλάδα, Ουκρανία, Βόρειος Αφρική. Ε, επίσης η τόσο αδύναμη και ασθενική μας οικονομία. Όλα αυτά έχουν προγραμματιστεί και έχουν ενταχθεί σε αυτό το προπολογισμό και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω που το κάνατε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Φερνάνδε. Προσωπικά θα ήθελα να σα ευχαριστήσω και το γεγονό πω έχετε χρηματοδοτήσει περισσότερο το Εράσμο και την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Είμαι νέο και γι' αυτό το κάνω. Είναι ε, προγράμματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και ελπίζω να ψηφίσουμε όλο και περισσότερου προπολογισμού τέτοιου είδου. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ συζητάμε θέματα προϋπολογισμού. Άρα λοιπόν θα πρέπει κάποια ουσιαστικά ζητήματα να τα συζητήσουμε. Ε, είναι αρκετά άρα για τα κονδύλια. Μπορούν να λύσουν τα ευρωπαϊκά προβλήματα. Νομίζω πως εν μέρη ναι. Αυτό το οποίο βρίσκω θετικό είναι πως για του χρόνου έχουμε προβλέψει περισσότερα χρήματα για επενδύσεις και καλωσορίζω το γεγονός πως για πρώτη φορά θα έχουμε περισσότερα κονδύλια για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης. Όμως, εδώ έχουμε μία πολύ σημαντική αδυναμία του προϋπολογισμού αυτού, που είναι το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ας μην ξεχνάμε πως ο κλάδος αυτός είναι ο κλάδος που δημιουργεί θέσεις εργασίας. Και αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που, αντιμετωπίζουμε. Χρειαζόμαστε ο κύριος Μαριάς, παρακαλώ, επόμενος ομιλητή. Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2016 που προβλέπει πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 153,5 δισεκατομμυρίων ευρώ ποσό που είναι ψίχουλα αν συγκριθεί με το 1,6 τρισεκατομμύρια ευρώ που διέθεσαν τα κράτη μέλη για να διασώσουν τις τράπεζες. είναι ψίχουλα αν συγκριθούν με το 1,1 τρισεκατομμύριο ευρώ που διαθέτει ο κύριος ντράγκη για την ποσοτική χαλάρωση και για την αγορά δημοσίου και ιδιωτικού χρέους όμως ακόμη και στο πλαίσιο αυτό της δημοσιονομικής λιτότητας του προϋπολογισμού του δύο πρέπει να διατεθούν τα κονδύλια αυτά κυρίως για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τη στήριξη των ανέργων για το χτύπημα της φτώχειας για την ενίσχυση της δράσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την κοινωνική οικονομική και εδαφική συνοχή της ένωσης για τη βιώσιμη γεωργία για την περιφερειακή ανάπτυξη ιδίως των νησιωτικών περιοχών.

δώσαμε την εντολή στην Επιτροπή για να επιτύχει. Αν θέλουμε και το Κοινοβούλιο να είναι επιτυχέ, είναι σαφές ότι, ότι πρέπει να επενδύσουμε στην οικονομία και στην οικονομική ανάπτυξη, γιατί αυτό θα είναι η απόδειξη της ε, ε, επιτυχημένης μας προσπάθεια. Είμαι πεπισμένος όσον αφορά την πολιτική συνοχής ε, ότι αυτή είναι ένα σημαντικός παράγοντας για πολλά κράτη-μέλη και τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι οι πολιτική συνοχής επιτρέπουν ε, σημαντικές επενδύσεις σε πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως το σχέδιο Juncker είναι και αυτό σημαντικό και θα πρέπει να είναι ε, ε, επιτυχές ε, θα πρέπει να είναι μια κοινή επιτυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι θα πρέπει να τονίσουμε την ε, στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο καθώς και για μικροπεριφερειακές στρατηγικές. Κυρία Μορβάη, τώρα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Σαν μουσική ακούστηκε στα αυτιά μου ότι ο προϋπολογισμός ε, της Ένωσης για το 2016 είναι κάτι που θα θα επιτρέψει να δοθεί βοήθεια στις στοχότερες χώρες και ότι θα υπάρξει ε, συνοχή και αλληλεγγύη ανάμεσα στις πλουσιότερες και τις φτωχότερες χώρες. Φυσικά μιλάμε κάπως γενικόλογα για όλα αυτά όπως ήθιστε. Γι' αυτό θα θέλουν και τον εισηγητή. Απτά μέτρα, τι ακριβώς θα γίνει δηλαδή για ποιες γραμμές μιλάμε στον προπολογισμό. Ας πούμε, ένας Ούγγρος πολίτης τι μπορεί να περιμένει όσον αφορά τις προσπάθειες εντό του πλαισίου του προπολογισμού ώστε να πάψει η οικονομική μετανάστευση από την Ουγγαρία προς άλλες χώρες της Ένωσης. Και πώς θα εξασφαλίσουμε τη βελτίωση των εισοδημάτων. Θα ήθελα λοιπόν συγκεκριμένες απαντήσεις. Ευχαριστώ. Και τώρα παρακαλώ την Επίτροπο να πάρει το λόγο, κύριε Γεωργίου. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους όσοι έλαβαν μέρος και συνέβαλαν στη συζήτηση. Θα προσπαθήσω να είμαστε το δυνατόν πιο συνεκτική και να δώσω απαντήσεις σε ερωτήσεις που ετυπώθηκαν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς, Ακούστηκε μια σειρά σχολείων για τη διαφορά, την απόκληση μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών για τον προπολογισμό του 2016 και ορισμένοι εξέφρασαν την ανησυχία ότι τα 10 δισεκατομμύρια στι αποκλήσει, ότι είναι περισσότερε δηλαδή αναλήψει υποχρεώσεων κατά 10 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια από τι πληρωμέ, θα μπορέσουμε να καλύψουμε το κενό το οποίο ιδιαίτερα χαρακτήρισε τον περσινό προπολογισμό. Εμεί όμω πιστεύουμε ότι δεν θα συμβεί αυτό. Για δύο λόγου. Πρώτον, λόγω των όλων ε, ιδιαίτερων μέτρων που λαμβάνουμε με το σχέδιο δαπανών που έχει ζητήσει και το Κοινοβούλιο ώστε να μειώσουμε από 24,7 στα 20 του εφέτος και του χρόνου στα 2 δισεκατομμύρια το ποσό των ανεξόφλητων λογαριασμών. Τα 2 δισεκατομμύρια είναι φυσιολογικό επίπεδο ανεξόφλητων λογαριασμών. Θα έχουμε μπει στην ομαλότητα δηλαδή. Δεύτερον, το 2016 τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι έχουμε ξεφύγει από την πίεση του προηγούμενου δημοσιονομικού πλαισίου, το οποίο επέρσι και εφέτος απαιτούσε σημαντικές πληρωμές, αλλά δεν έχουμε ακόμα μπει στην πίεση των πληρωμών του προσεχούς δημοσιονομικού πλαισίου. Άρα το 2016 είναι φυσιολογικό να έχουμε αναλήψει υποχρεώσεων περισσότερες σε ποσά από ότι οι πληρωμές, τα 10 δισεκατομμύρια αυτά τα οποία έχουμε υπολογίσει. Και σας ε, διαβεβαιώ ότι θα παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή κατά την εκτέλεση του προπολογισμού το κατά πόσον διαχειριζόμαστε σωστά τις πληρωμές ιδιαίτερως. Δεύτερον, ανησυχία εκφράστηκε ως προς τα οικονομικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τον υπολογισμό των ποσών που θα πρέπει να καταβληθούν για τη συνοχή. Ποια θα είναι, ποια θα είναι η πυρκοδότηση για τη συνοχή δηλαδή ανάλογα με τη χώρα, δεδομένου ότι υπάρχει μετακίνηση της, του επίπεδου των χωρών ανάλογα με το ΑΕΠ τους που τροποποιείται. Θα ξαναγίνει ο υπολογισμό λοιπόν το 2016 και αναλόγως θα επηρεαστεί και η πυρκοδότηση για την συνοχή. Επίσης, αρκετοί ομιλητές έθεσαν με έμφαση την ε, απέτηση ο προπολογισμό αυτό να είναι διαφορετικό, να είναι επικεντρωμένο περισσότερο σε προτεραιότητε, να είναι περισσότερο εστιασμένο, όπω είπε ο κ. Ε, στα αποτελέσματα, στην αποτελεσματικότητα, ή ότι θέλουμε να είναι ένα προπολογισμό ο οποίο θα διαχειρίζεται πολύ προσεκτικά την διοικητική πλευρά. Και όντω, προ αυτή την κατεύθυνση βαίνουμε κι εμεί. Είμαστε όμω σαν το ε, Queen Mary. Χρειάζεται χρόνο για να αλλάξει ρότο δηλαδή αλλά θα το πράξουμε και θα το δείτε σε το χρόνο. Ότι χρειάζεται χρόνος, αλλά χρειάζεται και να δούμε τους, τα πολλαπλά ωφέλη από τις επενδύσεις. Επενδύσεις φερειπίν στη συγκαιροτομία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Βεβαίως θα το κάνουμε και από εκεί θα προκύψει και η απασχόληση. Από εκεί θα δούμε την βελτίωση των προϋποθέσεων διαβίωσης σε χώρες όπου παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας και βέβαια στο σχεδιασμό του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνουμε όχι μόνο τις δαπάνες μας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το κόσμο επί παραδείγματι, αλλά και τον τρόπο, τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται όλα αυτά με το επενδυτικό σχέδιο Juncker για να είναι πιο αποτελεσματικό. Συγκεκριμένα ρωτήσατε για την Ουγγαρία. Τι μπορεί να προκύψει για τους πολίτες Ουγγαρίας σαν αποτέλεσμα του προϋπολογισμού. Κοιτάξτε, προφανώ δεν πρέπει να το ξανασυζητήσουμε με τα λεπτομερέστερα στοιχεία όταν, έχει όρθα, όταν έρθει η ώρα. Τώρα δεν έχω επαρκή χρόνο για να το αναλύσω. Αλλά θα δείτε ότι ο προπολογισμό του 2016 διαφέρει σε σχέση με του προηγούμενου. Πώ ότι θα υπάρχει σαφής διάσταση συνοχής διαφορετικά ταμεία και γεωργίας από το Γεωργικό Ταμείο για την Ουγγαρία γιατί έχει, έχει μεγάλο κομμάτι η γεωργίας οικονομία της ε, Ουγγαρίας αλλά ταυτόχρονα ελπίζω θα μπορέσουμε να δούμε και κομμάτι από το σχέδιο Juncker χρήματα δηλαδή τα οποία θα επενδυθούν για να αφυπνίσουν την ε, ενυπνώση ρευστότητα που υπάρχει και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε την απάντηση και νομίζω ότι εγώ θα μπορούσα να δώσω την απάντηση στον έρθει η ώρα για το τι βλέπω σαν ε, όφελος από τον προβολισμό αυτό εάν ήμουν Ουγγαρέζα. Και κύριε Φερνάντες, είμαστε στη διάθεσή σας μέρα νύχτα, προτιμάμε βέβαια μέρα, αλλά όποτε θέλετε με διστάστε. ευχαριστώ. πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Φερνάντες. Σας, Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την συνεργασία της και για την θετική της στάση. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην ε, οικοδόμηση ε, του προϋπολογισμού για το 2016 σε αυτή την εντολή μέσω του Τριλόγου. Βέβαια, ε, στην, ε, στην Επιτροπή πιστεύουμε ότι είμαστε συνεπείς, φιλόδοξοι, αλλά και αυστηροί και ελπίζω πως και το Συμβούλιο θα έχει την ίδια στάση. Ελπίζω συνοχή από πλευράς του Συμβουλίου και πέρα από αυτό Ξέρουμε όλοι πως για να εγκριθεί το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ε, ανάγκη να συνανοηθούμε και έπειτα τα κάτι μέλη να καταψηφίζουν προπολογισμού τους οποίους, ε, οι οποίοι συμφωνούν με το ίδιο το PDP το οποίο εκείνα ενέκριναν και μάλιστα και κάτω από αυτό το ίδιο το πολιετές ε, δεν είναι αυτό συνοχή δυστυχώς. Υπάρχουν κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που Κατά εξακολούθηση καταψηφίζουν τους προϋπολογισμούς και λένε μάλιστα στην κοινή γνώμη δεν ε, γίνεται αυτό γνωστό. Εμείς από την πλευρά μας λέμε ότι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας. Θέλουμε ευελιξία και αυτό λόγω της ευελιξίας ακριβώς εγκρίναμε το πολιετές πλαίσιο για το 2014-2020 που είναι μικρότερο από αυτό το 2007 και 2013. Ευελιξία σημαίνει να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα της ευελιξίας και ε, περιθώρια που παλαιότερα δεν είχαν, τα αποθεματικά τα οποία δεν είχαν χρησιμοποιηθεί και θα τα χρειαστούμε για να μπορέσουμε να τηρήσουμε τους στόχους, να πετύχουμε τους στόχους που θεσπίσαμε σε σχέση με το 2020. Αλλά θα εξακολουθήσουμε να ελαχιστοποιούμε όσο γίνεται τον αντίκτυπο που έχει ε, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων σε αυτά τα προγράμματα. Πιστεύω πως συμφωνούμε με το στόχο ανάπτυξη, απασχόληση, εσωτερική αλληλεγγύη, εξωτερική αλληλεγγύη, ασφάλεια και γι' αυτό και ελπίζω ότι θα είναι μαζική η ψήφος υπέρ αυτής της έκθεσης και της εντολής. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Και τώρα Ολοκληρώνεται η συζήτηση αυτή και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Πριν να δώσω τη θέση μου στην κυρία Γιατρεμάκη, έχω να κάνω μία ε, ανακοίνωση. Σύμφωνα με το άρθρο 190 παράγραφος 1, η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου με ενημέρωσε ότι αύριο Κατά την έναρξη της συζήτησης σε σχέση με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, θα ζητήσει την αναβολή της εν λόγω συζήτησης, έτσι ώστε να είναι παρούσα και η ύπατη εκπρόσωπος. Ευχαριστώ.